Session. Κυρίσω την επανάληψη της ε, Συνόδου. Τα πρακτικά της χθεσινής συναριάσεων ε, είναι στη διάθεσή σας. Ε, εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, σχόλια, τα θεωρούμε εγκεκριμένα και να περάσουμε στο πρώτο σημείο της απογευματινής μας συνεδρίασης που πρόκειται για την κοινή συζήτηση σχετικά με την φάρμα